Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzungen vom 9. Τα πρακτικά της 9ης και 10ης Μαΐου του 2012 είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνονται τα πρακτικά